τελειώσει. Ούτε καν όταν θα υιοθετηθεί αυτό το κείμενο και υπογραφή. Τότε θα αρχίσει η εργασία μάλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Εκ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψήφιση, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Περνάμε αμέσως στο ακόλουθο σημείο στην ημερησία διάταξη. Θέλω να σας επαναλάβω εδώ κάτι. Ότι υποτίθεται ότι θα ολοκληρώσουμε στις 12 τα μεσάνυχτα σε σχέση με τις 12 τα μεσάνυχτα πέρα από αυτό το όριο περιπλέκονται τα θέματα με θέματα διερμηνίας όχι μόνο για απόψε αλλά και για αύριο. Γι' αυτό παρακαλώ λοιπόν θερμά να είσαστε το δυνατόν συντομότερη στις παρεμβάσεις σας. Να εφαρμόζουμε το χρονικό όριο με μια λογική οικονομική διαχείριση προσαρμοζόμενη στον χρόνο αγορητών. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του κυρίου συναδέλφου Κουέλιο για την εφαρμογή των διατάξεων και εκτιμένου του Σέγγεν στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία. Θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος κύριος Κάρλος Κοέλιο, ο συζητητής. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ στα Ισπανικά, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στα Πορτογαλικά ο μιλητή, κύριε Επίτροπε Μάνστρομ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα θεμελιώδη σημεία. Πρώτον, για την διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 όταν εντάχθηκαν η Ρουμανία και η Βουλγαρία προσπάθησαν να ενταχθούν πλήρως στον χώρο Σέγγεν. Για να μπορέσει το Συμβούλιο να λάβει απόφαση όσον αφορά τα εσωτερικά αυτά θέματα είναι αναγκαίο οι διαδικασίε αξιολόγηση να πιστοποιήσουν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις και όρους για την εφαρμογή των σημαντικών θεμάτων του κοινοτικού κεκτημένου. Προστασία δεδομένων, σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, τα εναέρια σύνορα, τα χερσαία σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, την ε, αστυνομική συνεργασία και τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Οι αξιολογήσεις αυτές ξεκίνησαν όσον αφορά την προστασία δεδομένων πρώτα. Θέλαμε να επιστοποιήσουμε ότι κάθε ένα από αυτά τα κράτη-μέλη ήταν επαρκώς προετοιμασμένο για να υλοποιήσει όλες τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουν αποκτηθεί είναι προηγούμενος όρος και προϋπόθεση για το σύστημα πληροφόρησης Schengen που θα δίνει τη δυνατότητα της μεταφοράς αυτών των στοιχείων σε αυτές τις χώρες. Με αυτή την απόφαση γίνεται ένα πρώτο βήμα λοιπόν όσον αφορά την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και των άλλων χωρών και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Επίσης, σε σχέση με τα άλλα στοιχεία σε σχέση με την λήψη απόφασης ε, δεν είχαν αποσταλεί τα ε, στοιχεία αξιολόγησης, τα follow-ups ε, που θα είχαν δώσει δυνατότητα στο Ευρωκοινοβούλιο να έχει όλες τις αναγκαίες ε, πληροφορίες για την εκπόνηση αυτών των στοιχείων. Μόνο μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου παραδόθηκαν, δόθηκαν αυτά τα στοιχεία από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ για την προσπάθεια του πρέσβεως ε, της Ρουμανίας να εξευρεθεί λύση, ώστε αυτή η κατάσταση να ε, αντιμετωπιστεί όπως έπρεπε και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Μέσω διαβαθμισμένων εγγράφων τα οποία μπόρεσαν να διαβιβαστούν αυτό έδωσε τη δυνατότητα να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε όμω το ίδιο πρόβλημα. Όταν έρχεται η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τι άλλε πτυχέ ε, του κεκτημένου του Σέγγεν, θα πρέπει το δυνατόν γοργότερα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων. Τρίτο, όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση Ρουμανία και Βουλγαρία. Ε, σε σχέση με τη Βουλγαρία υπήρξαν κάποιε ελλείψει που διατυπώθηκαν ε, όσον αφορά την υλοποίηση του, οδηγίας του Συμβουλίου της, ε, της Ευρώπης και βρέθηκαν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων εν τέλει. Η Βουλγαρία έδωσε αναγκαία προσοχή στην παρακολούθηση αυτών των θεμάτων και το Συμβούλιο συνεπέρανε ότι οι αναγκαίες αυτές ε, προϋποθέσεις ήταν πλέον διασφαλισμένες στην ε, Ρουμανία σε σχέση με αδυναμίες όσον αφορά ε, νομοθετήματα καθώς επίσης ε, και την διαδικασία προστασίας δεδομένων καθώς επίσης και τις περιοδικές εκθέσεις ή ελέγχους για το κεκτημένο. Έτσι λοιπόν αυτά τα οποία απομένουν δεν παρακολύουν η χώρα αυτή να εφαρμόζει με αποτελεσματικότητα όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία των δεδομένων. Έτσι λοιπόν υλοποιούνται οι συνθήκες και οι όροι ώστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να μπορέσουν να ενταχθούν στο κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά το μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ανάγκη το δυνατόν γοργότερα να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ευρωπαϊκής αξιολόγησης που θα είναι απλός, θα είναι αποτελεσματικός και διαφανής όσον αφορά το, τη ζώνη Σέγγεν απέρριψε τις προτάσεις που του υπευλήθησαν το Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο Οκτώβριο. Και έτσι θα πρέπει να αναλυθεί το δικαίωμα ιδίας πρωτοβουλίας των δυνατόν ταχύτερα όσον αφορά την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Θα λάβει τώρα τον λόγο η Επίτροπος Μάλμστρομ για να παρουσιάσει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά. Thank you, Mr. President. Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κοέλιο, κυρίες και κύριοι, ε, Έχω την υπεποίθηση ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ώστε να έρθουν ε, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μέχρι το 2011 και η Κομισιόν θα υποστηρίξει πλήρω αυτέ τι δύο χώρε για να περάσουν την αξιολόγηση Σέγγεν. Είναι ευθύνη του Συμβουλίου να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση για το Σέγγεν και με βάση τι αξιολογήσει αυτέ το Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα έρθουν ή όχι οι εσωτερικοί έλεγχοι βρίσκονται να εξελίξει αυτέ οι αξιολογήσεις, άρα είναι πολύ νωρί για να πούμε το οτιδήποτε. Τα πρώτα βήματα όμως στέφθηκαν ε, με επιτυχία, ε, σχετικά δηλαδή με την προστασία των δεδομένων, πράγμα το οποίο ε, επιτρέπει τώρα στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία να έχουν πρόσβαση στο ΣΥΣ, στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα πρέπει να ενημερώνουν το ε, Κοινοβούλιο ε, σχετικά με τις αξιολογίες αυτές. Τα κράτη-μέλη ε, θα υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί το, η αξιολόγηση είναι ευθύνη του Συμβουλίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Και έτσι λοιπόν ε, δέχομαι την πρότασή σας και το φθινόπωρο θα ε, προτείνω ε, ένα νέο μηχανισμό αξιολόγησης μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Αβώνα για του λόγου που αναφέρεται κύριε Κοέλου. Και νομίζω ότι και τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό. Τα κράτη-μέλη, βέβαια, ε, θα πρέπει να συμμετέχουν για να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του ότι θα, θα εφαρμοστούν όλα τα συνοδευτικά μέτρα που είναι προπόθεση για την άρση ε, των ιστορικών ελέγχων, αλλά και για του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και την πολιτική θεωρήσεων. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και αυτό να είναι πλήρω ενημερωμένο για τα αποτελέσματα αυτή τη αξιολόγηση. Και γι' αυτό η Κομισιόν ε, προτείνει να καλυφθούν οι σημερινές αδυναμίες όπως ε, ε, προτείνει και η έκθεση που συζητάμε. Χρειάζεται η υποστήριξη του Κοινοβουλίου που θα είναι πολύτιμη στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ με την πρακτική 10 δευτερόλεπτα να αφαιρείτε το μικρόφωνο ήταν ο μόνος τρόπος να καταλήξουμε σε αυτή την καταληκτική προθεσμία τώρα. Και εξ ονόματος του ΕΛΚΑ 1,5 λεπτό η κυρία Νέντερτσέβα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο για την έκθεση πρόοδου. Ε, με βάση τα θετικά αποτελέσματα ε, από του ελέγχου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, είναι δυνατό να οριστεί μια ημερομηνία κατά την οποία το ΣΥΣ θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην ε, Βουλγαρία. Όσον αφορά την πρόσβαση, την ε, ένταξη τη Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόσβαση τη χώρα στο ΣΥΣ, αυτό προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό σε όλου του κατοίκου τη χώρα, διότι αυτό θα οδηγήσει στην άρση των ελέγχων στα σύνορα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της ε, σημερινής κυβέρνησης της Βουλγαρίας που ε, κάλυψε τα κενά ε, και τις αδυναμίες του παρελθόντος. Ο χώρος Σέγγεν δεν σημαίνει μόνο ελευθερία κίνησης, αλλά σημαίνει και ισχυρότερη τελωνιακή ε, συνεργασία, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων και το λαθρεμπόριο. Η πρόσβαση της Βουλγαρίας στο Σέγγεν είναι μέρος του ονείρου της Βουλγαρίας για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που έχουν γίνει. Το follow-up ε, είναι η εγγύηση ότι ο υποδομητικός διάλογος θα συνεχιστεί μεταξύ όλων ημών. Ε, αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι μια πραγματικότητα στη Ρουμανία και στην Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ένσιο, δύο λεπτά εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χθε γιορτάσαμε την 25η επέτειο ε, του ε, της Ευρώπης ε, με μια κινητικότητα χωρίς σύνορα. Και η Επίτροπος δήλωσε ότι αυτή η ελευθερία κίνησης είναι πραγματικά το πιο σημαντικό ε, σύμβολο ε, αυτής της Ευρώπης για τους πολίτες της. Ε, το Σέγγεν είναι μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 30 χρόνια. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Σέγγεν, χρόνια πολλά στην ελευθερία κίνησης και στην κατάργηση των ελέγχων που συζητάμε σήμερα. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες είναι πραγματικά έτοιμες να αποδείξουν ότι είναι ικανές να ε, μπουν στο σύστημα Σέγγεν. Και αυτό προς όφελος των πολιτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αλλά και προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών για μια πραγματική Ευρώπη χωρίς σύνορα. Μια οικονομική και κοινωνική Ευρώπη. Βεβαίως τα δύο αυτά κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, σεβαστούν τον οδικό χάρτη που έχει χαράξει η Κομισιόν και είναι πολύ καλό που το Κοινοβούλιο ε, επέτυχε να διαδραματίσει τον ρόλο του ως θεματοφύλακα των δικαιωμάτων ε, μέσα σε ένα μοντέλο διαφάνειας και συνεργασίας ε, στα πλαίσια μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς το συμφέρον όλων. Αλλά ας είμαστε σαφείς για ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ε, έχει άλλο μέλημα παρά ε, την, ε, να είναι στην υπηρεσία των πολιτών με μεγαλύτερη ισότητα και ελευθερία κίνηση στην Ευρώπη. Υποστηρίζουμε λοιπόν τον κύριο Κόελιο. Αφαιρέθηκε το μικρόφωνο. Θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Η κυρία Γκρίσμπεκ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν μερικές μέρες με τον πρόεδρο Μπούζεκ και Μπαρόζο γιορτάσαμε την επέτειο των συμφωνιών Σέγγεν και σήμερα θέτουμε ένα νέο λιθάρι απόψε το βράδυ αργά περνούμε από τον προβληματισμό στην δράση και στην συνεργασία προϋποθέσεις απαραίτητες οι οποίες είναι αυτές της κατάργησης των ελέγχων στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Ρουμανία που πληρούν σιγά σιγά τις προϋποθέσεις για τις πρώτες αξιολογήσεις. Οι δύο αυτές οι χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν την προστασία ε, των ε, προσωπικών δεδομένων και αυτό ε, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση των δύο αυτών χωρών και θα επιτρέψει την επιμερία όχι μόνο για αυτές τις χώρες αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τα ρεύματα παράνομης μετανάστευσης, διεθνούς εγκληματικότητας και άλλες μάστιγες θα δύο ε, παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Αφαιρέθηκε το μικρόφωνο. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ένα λεπτό η κυρία Σντανόκα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κυρία Επίτροπε, εφόσον το ΣΥΣ είναι αναπόσπαστο μέρος ε, ε, του συστήματος Σέγγεν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Είμαι από νέο κράτος μέλος και θυμάμαι πώς η Λετωνία ήθελε να προσχωρήσει στην περιοχή. Γι' αυτό χαιρετίζω την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα. Από την άποψη αυτή η ομάδα μου συμμερίζεται την άποψη της του εισηγητή ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πώς τα προβλήματα ρυθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες μας για την προστασία των δεδομένων. Θα ελπίζω επίσης ότι ε, ε, ε, η ανεπάρκεια των χρονοθυρίδων δεν θα είναι σημαντικό εμπόδιο. Σημεριζόμαστε τις ανησυχίες για την αξιολόγηση του νέου μηχανισμού Σέγγεν. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ασκήσει έλεγχο δημοκρατικό και χαιρετίζω την δήλωση της κυρίας Μάλστρομ ότι αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ. Ισπανικά έχει. Όχι, είχε γαλλικά μόνο. Δεν λειτουργεί η διερμηνία. Υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη διερμηνία. Ε, Μπορείτε να επανέλθετε και να ξαναξεκινήσετε παρακαλώ. Τώρα, τώρα, τώρα παρακαλώ. Μπορείτε να ξαναξεκινήσετε τώρα την παρέμβασή σας παρακαλώ. Yes, yes. Okay. Έχετε τον λόγο. Ξεκινήστε παρακαλώ. Ρωμανία και η Βουλγαρία έχουν υιοθετήσει τις κοινοτικές οδηγίες 2007 και σήμερα συζητούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κεκτημένο κοινο, ε, το κοινοτικό που υιοθετήθηκε από τα δύο τελευταία μέλη. Είναι από τα τελικά βήματα προς την προσχώρηση για την εξάλληψη των διασυνοριακών ελέγχων στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Η εξολόγηση ήταν θετική σχετικά με την εξάλληψη των συνοριακών ελέγχων και ορισμένες, ορισμένα μειονεκτήματα και ανεπάρκειες θα έπρεπε να εξαλειφθούν σύντομα. Ελπίζουμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία τεχνικά θα ε, είναι έτοιμες για το ΣΥΣ 2 πριν από τον Οκτώβριο 2010 σύμφωνα με τον χάρτη πορείας. Χάρη σε αυτό θα μπορεί να ανοιχθεί το σύστημα Schengen σε δύο κράτη-μέλη με την ε, δέουσα προσοχή και προστασία των πολιτών. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Την Πρόεδρος, θα λάβει τώρα εξ ονόματος της Ευρώπης Ελευθεριών και Δημοκρατίας για τρία λεπτά ο κύριος Δάφτον, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, το Σέγγεν ήταν ένα αντάλλαγμα για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση ατόμων ε, και μέτρα για την ασφάλεια και προστασία παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέρος του Σέγγεν, του κεκτημένου Σέγγεν, ε, συμμετέχουμε στο σύστημα καταπολέμησης του εγκλήματος. Το κεκτημένο επίσης δίνει μια ευρύτερη πλατφόρμα ε, για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα μετά την προσχώρηση στο ΣΥΣ της Βουλγαρίας και Ρουμανίας το βασικό θέμα είναι αν τα θέματα αυτά, τα, οι χώρες αυτές μπορούν να εγγυηθούν επίπεδο ελέγχου για την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ήπειρο υπήρξε αντίθεση στο να περάσουμε σε δεύτερη εξέλιξη του συστήματος στο Σέγγεν. Η ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος ε, τέθηκε επιτάπητος. Εμείς έχουμε ανεξάρτητους ελέγχους και δεν ε, συμμετέχουμε ε, σε ταξίδια χωρίς θεωρήσεις πρέπει να μετριάσουμε την αύξηση της εγκληματικότητας που θα είναι συνέπεια του ανοίγματο του συνέρων. Το Σέγγεν έχει αυξήσει την δυνατότητα λαθρεμπορίας, λαθρέας διακίνησης. Ε, πρέπει να βασίζεται η ελευθερία πάνω στην εμπιστοσύνη και την ικανότητα των κρατών μελών να ε, ε, ασκούν ελέγχου σε κατάλληλο επίπεδο. Η επέκταση του ΣΥΣ αυξάνει το παράθυρο διαφθοράς και επιτρέπει επίσης την, εγκληματίε να μπαίνουν στο σύστημα, να κάνουν hacking. Ίσως χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για το σύστημα Schengen κυρίως με το ΣΥΣ2 παραδείγματος χάρη σε ένα σημείο εκεί όπου έχουμε αποθήκευση βιομετρικών στοιχείων. Πρέπει να υπάρχει προστασία. Επίσης το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές απόψεις. Μπορεί να υπάρχει κακή χρήση των στοιχείων με αυξανόμενο αριθμό χωρών που, που μπαίνουν στο σύστημα, στο κεκτημένο, ο κίνδυνος αυξάνεται, διότι έχουμε πρόσβαση στο ΣΥΣ. Δεν ξέρουμε πόσο ανταλογισμικά αυτά είναι ασφαλή. Ε, έχουμε επίσης θύματα, θύματα ιών. Όσο ευρύτερο είναι το σύστημα, όσο περισσότερα είναι τα στοιχεία στα οποία υπάρχει πρόσβαση και τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα κατάχρησης θα πρέπει να υπάρχει προχωρημένη ασφάλεια και ακόμα με τις καλύτερες προθέσεις δεν υπάρχει προστασία από τον κίνδυνο παραβίασης του συστήματος. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τώρα αυτόν τον γύρο αγοριτών. Περνάμε στον γύρο Catch the Eye. Έχουμε πέντε συναδέλφους που πρόσεξα και έχω εγγράψει. Πρώτα απ' όλα, για ένα λεπτό, η κυρία Αντωνέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητικό Έλιο για τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε με το φάκελο αυτό και να το συγχαρώ για την εργασία του. Υποστηρίζω τα όσα δήλωσε πριν από λίγα λεπτά, όχι μόνο σχετικά με την αξιολόγηση, σχετικά με την προστασία των δεδομένων, αλλά και για τους άλλους τομείς οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν. Το Συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει τη διαθέτηση ε, τις, όλες ε, τις πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στο Ευρωκοινοβούλιο του ώστε αυτό να μπορεί να λάβει την κατάλληλη απόφαση. Ελπίζω να μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση γνωρίζοντας ε, όλα τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Βατσέσκου τώρα παρακαλώ. Η κυρία Μπατσέσκου έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο ε, που ασχολήθηκε με μια σημαντική εισήγηση για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Θέλω να πω ότι στη Ρουμανία υπάρχει ένας νόμος ο οποίος υιοθετήθηκε τώρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι μια πρόοδος για τη χώρα μας η οποία θέλει να προσχωρήσει στο χώρο Σέγγεν. Το Υπουργείο έχει επιτελέσει πρόοδους πρόσφατα και θα έχουμε στο 2011 στοιχεία στα φέστερα σχετικά με τα μέτρα που θα έχουν ληφθεί σχετικά ακόμα και με το θαλάσσιο σύστημα το ναυτικό ΣΥΚΟΜΑΡ. Με αυτήν την μεταρρύθμιση θα δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τη Frontex και με άλλους οργανισμούς για την επιτήρηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπασέσκου. Θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Λούχαν Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Κοέλιο. Πράγματι έκανε εξαιρετική δουλειά για την Ρουμανία και την Βουλγαρία. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Ρουμανία είναι πραγματικά ένα υπόδειγμα καλής πρακτικής όσον αφορά την ασφάλεια ε, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Και η Ρουμανία όπως και η Βουλγαρία πληρεί τις προϋποθέσεις για να έχει πρόσβαση στο σύστημα ΣΥΣ. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και η Κομισιόν θα πρέπει να ε, υποστηρίξει τις δύο χώρες ούτως ώστε να ε, έχουν αίσιο πέρας και οι άλλες αξιολογήσεις και να έχουν πρόσβαση στον ε, κοινό αυτό ευρωπαϊκό χώρο. Πρόκειται για μια διεύρυνση που βασίζεται στις... Σας ευχαριστώ. Κύριο Σικέσκη, παρακαλώ έχει τον λόγο. What... Σας ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι εποφελούνται από το σύστημα SIS που καθιστά εφικτή την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την ε, κυκλοφορία των αγαθών. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνεται αυτό όμως καθημερινά είναι σημαντικό να υπάρχουν οι τεχνικές, τεχνολογικές υποδομές για την εποπτεία αυτών των διεργασιών. Γνωρίζω από προσωπικά βιώματα και πείρα ότι το έργο χωρών που εντάσσονται στο Σέγγεν είναι κυρίως η υλοποίηση των και του κεκτημένου και των υποχρεώσεών τους. Είναι προς όφελος, προς το κοινό όφελος ε, και προς όφελος της ασφάλειας και πρέπει να γίνονται δεκτές προδιαγραφές και διατάξεις. Πρόεδρος, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση του κυρίου Μπόης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, λέει ο κύριος Μπόρης, να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο που είναι επαΐων στα θέματα Σέγγεν και έχει κάνει τεράστιο έργο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι αξιολογήθηκαν θετικά η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχουν άρει όλα τα προβλήματα αυτές οι δύο χώρες για να προχωρήσουν στην επίτευξη θετικών ε, αποτελεσματών ως έκβαση. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι πολύ σημαντική εδώ. Είναι η σημαντικότερη. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σε σχέση και με τα βιομετρικά στοιχεία στο μέλλον, αλλά μην ξεχνάμε ότι αναμένει αυτή η διεργασία την προσοχή που πρέπει για να προαχθούν αυτά τα θέματα. Εύχομαι στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία το ίδιο που ζήσαμε σε σχέση και με τους ε, Τσέχους, ε, όταν, Τσέχους αδερφούς όταν ξεπεράσαμε τα ιστορικά σύνορα. Αυτό αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη αυτών των δύο χωρών. Ελπίζω ότι αυτές οι δύο χώρες θα υλοποιήσουν όλες τις ε, διατάξεις και προϋποθέσεις και εύχομαι κάθε επιτυχία. Πρόεδρος, η κυρία Μάλμστρομ για να τοποθετηθεί σε σχέση με τις παρεμβάσεις των διαφόρων αγοριτών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω πολλά να πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συνένεση ε, και όντως ε, είχαμε ένα λόγο να γιορτάσουμε αυτή την εβδομάδα για το Σέγγεν που είναι ένα επίτευγμα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Ε, αντιπροσωπεύει την ελεύθερη κυκλοφορία σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Ε, και ο, ο χώρος ε, Σέγγεν θα ενισχυθεί με δύο νέα μέλη πολύ σύντομα. Προς το παρόν η πρόσβαση βέβαια στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Χρειάζεται ακόμα να γίνει κάποια δουλειά στις ε, χώρες αυτές για την αστυνομική συνεργασία, παραδείγματος χάρη την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και φυσικά χρειάζεται ε, πολύ προσεκτικό monitoring. Ε, μέχρι το τέλος της χρονιάς σκοπεύω εγώ προσωπικά να επισκεφτώ τις δύο χώρες για να δείξω την υποστήριξή μου και να μελετήσω επιτόπου την πρόοδό τους. Και θέλω να ευχαριστήσω τις δύο χώρες για την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Η εμπιστοσύνη φυσικά είναι πολύ σημαντική και για τα άλλα κράτη-μέλη για να, για να δουν συγκεκριμένα αποτέλεσμα αποτελέσματα, ώστε να έχουμε ένα αίσιο τέλος σε αυτή την ιστορία και βεβαίως για να βελτιωθεί και να αυξηθεί η διαφάνεια του συστήματος και για να αυξηθεί και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση και την εφαρμογή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και γι' αυτό ελπίζω ότι από κοινού μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό, για αυτό το νέο μηχανισμό αξιολόγηση. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για τη δουλειά που έκανε για αυτέ τι δύο χώρε και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία μαζί μα. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με παρέμβαση του εισηγητού κυρίου Κουέλιο, που τον συγχαίρουμε ήδη και έχει δύο λεπτά για την παρέμβασή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τέσσερι τελικέ παρατηρήσει. Πρώτον, για να ευχαριστήσω τις, ε, την κατανόηση και την, ε, τους των συναδέλφων και ευχαριστώ για την καλή συνεργασία του σκιώδης εισηγητές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω δεύτερον ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση για αυτές τις πρωτοβουλίε. αλλά επίση να ζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται σε προθεσμία έξι μηνών όσον αφορά την παρακολούθηση που θα δίνονται σε σχέση με τις ε, ε, συστάσεις που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Τρίτον, να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα που κάνουμε. Υπάρχουν άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, όπως ε, η κυρία Επίτροπος Μάνστρομ υπενθύμησε πολύ καλά μόλις πριν από λίγο. Τέταρτον και τελευταίο, θέλω να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο Μάνστρομ για τι εγγυήσει, τα ηχέγγυα που μα έδωσε ότι το φθινόπωρο θα υποβάλει μια πρόταση ιδίας πρωτοβουλία, νομοθετική πρόταση για το σύστημα αξιολόγηση. Αυτέ οι δύο χώρε αξιολογούνται αποκλειστικά μόνο από το Συμβούλιο. Εμεί χρειαζόμαστε όμω ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγηση, όπω είπε η κυρία Επίτροπο, που θα εμπλέκει όλες ε, τις, ε, όλα τα θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, αλλά επίση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίω ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγηση, το οποίο δεν θα στηρίζεται μόνο σε δύο προδιαγραφές και διατάξεις. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από κράτη που βρίσκονται εκτός και θέλουν να ενταχθούν στο Σέγγεν ένα κριτήριο αξιολόγησης πιο αυστηρό από εκείνο το κριτήριο το οποίο εφαρμόζουμε στα κράτη τα οποία βρίσκονται ήδη εντός Σέγγεν όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν και όλοι όσοι βρίσκονται ήδη στο σύστημα αυτό πρέπει να αποδείξουν αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Σέγγεν. Και οι καλύτεροι έλεγχοι πρέπει να υπάρχουν στα εξωτερικά σύνορα. Μόνο έτσι μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ασφάλεια του χώρου αυτού κυκλοφορία Σέγγεν. Να δώσουμε χέγγια στου πολίτε μα ότι μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε, λέει ο πρόεδρο. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά σα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι και το τελευταίο απόψε και που είναι η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με θέματα αθλητισμού, ιδιαίτερα